Θα, θα στο δείξω στην πράξη, θα βάζεις Thank you. Uh, Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε αυτήν την ε, μεικτή συνεδρίαση, κοινή συνεδρίαση που κάνουμε. Και πριν περάσω στην εμερήσια διάταξη, ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι διαθέτουμε την ερμηνεία σε όλες τις γλώσσες πλην της δανικής και μαλτεζικής. Και τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω την δόκτωρα Σαρούς Μιντήρο, αναπληρώτρια γραμματέα, Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει ήδη επισκεφθεί εμάς, το Κοινοβούλιο, και στο παρελθόν, άλλες δύο φορές, αυτή είναι η τρίτη φορά που έρχεται, επί τη ευκαιρία της ε, θέσης ε, ε, λειτουργία, της παρουσίασης καλύτερα, της ε, Έκθεση για την συνεργασία ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εταιρική σχέση. Η δόκτωρα Σάρο Σεμιγκύρο έχει ε, κάνει το μάστερ στη και τη, διδακτορική της ατριβή στα νομικά θέματα. Έχει βέβαια κάνει ασκήσει το δικαίωμα του δικηγόρου. Στη συνέχεια ασχολήθηκε σε πολιτικά ε, καθήκοντα ως υπουργό, ε, δύο φορές στη χώρα της και στη συνέχεια ε, ανέλαβε ως τρίτη αναπληρώτρια γενική γραμματέας για τη θέση του, γενικού, αναπληρωτή γενικού γραμματέα που θεσπίστηκε το 1997. Είναι η τρίτη λοιπόν που κάθε στο θόκο του αναπληρωτή γενικού γραμματέα. Και επίση θα πω ότι οι υποεπιτροπές μας θα πάνε στη Νέα Υόρκη στα μέσα Νοεμβρίου Ίσως γνωρίζετε ήδη ότι η ευκαιρία αυτή θα είναι χρυσή για την συνέχιση του διαλόγου που θα ξεκινήσουμε σήμερα μαζί σας και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να προαγάγουμε ακόμη περισσότερο τα θέματα των Ηνωμένων Εθνών στο Κοινοβούλιο με την ευκαιρία αυτή και να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε επίπεδο των επιτροπών και υποεπιτροπών μα ε, σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντο. Όπω είπα, είναι κοινή συνεδρίαση από την Επιτροπή Περιβάλλοντο, ε, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων, αλλά και Ισότητα των Φίλων, που είναι εδώ παρόντες μαζί με την Επιτροπή των Εξωτερικών και χαιρετίζω την παρουσία των ε, συναδέλφων μας εδώ. Ξέρετε ότι η ευκαιρία να ε, εξάρουμε τη συνεργασία μεταξύ ΗΕ και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται ποτέ. Είναι η τέταρτη φορά που ε, έχουμε την έκθεση αυτή που αποτελεί πολύ σημαντική ευκαιρία να εξάρουμε τη συνεργασία μας και αποτελεί μια ε, σαφή ένδειξη της δυνάμωσης εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων μας η έκθεση αυτή. Και χωρίς να χάσουμε περισσότερο χρόνο θα ήθελα να παρακολουθήσω τη δόκτωρα Ανιγκύρο να λάβει το λόγο, να κάνει την ε, παρουσίασή της και μετά η συνάδελφος κυρία Ζούλη θα αναλάβει την Προεδρία για να ακούσουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Προβλέπετε η συνεδρίασή μας να τελειώσει κάπου στις 7. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τους πάντες να είναι πολύ σύντομοι Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζούλη, Πρόεδρε τη Επιτροπής Ανάπτυξης, κύριε του Αντιπρόεδρε τη Επιτροπής των Εξωτερικών, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και ο κύριος Πάσο, η επίσκεψή μου είναι η τρίτη επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ανάπτυξη των κρατικών των αναπληρώτρια Γενικού Γραμματέως το 2007 και θεωρώ πολύ ευπρόσδεκτη αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα των επιτροπών μας σε σχέση με τους αλληλοσυνδεόμενους πυλώνες του έργου των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή την ανάπτυξη, την ειρήνη, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θέλω επί τη ευκαιρία να ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους πρόεδρους της Επιτροπής, αλλά και τους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι εδώ παρόντες από διάφορες επιτροπές σήμερα που ασχολούνται με θέματα των Ηνωμένων Εθνών, περιβάλλον, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα των φύλων και δημοσιονομικό έλεγχο. ότι, κυρίε και κύριοι, η Ευρώπη ανέκαθεν προσπιζόταν ε, τις, ε, την, ε, σε διεθνές επίπεδο επίλυση των διεθνών προβλημάτων και πάντοτε βοηθούσε στην ανέβριση κατάλληλης λύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαναλημμένως δηλώσει την δέσμευσή της, τη στράτευσή της, την ανοικοδόμηση ενός αποτελεσματικού πολυμερούς πλαισίου με ισχυρά Ηνωμένα Έθνη. Πολιτικά ισχυρά, και οικονομικά ισχυρά. Η οικονομική κρίση σήμερα επηρεάζει τις χώρες σας, τις ε, ιδιαίτερα στις πατρίδας ε, βαθιά και σημαίνει ακόμη περισσότερες ε, ακόμη περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδιόμενες χώρες στην εγκύτερη περιοχή της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαίνει ότι είναι λιγότερες, λιγότερες ζήτηση για εξαγωγές και ε, χαμηλότερες οι τιμές των βασικών προϊόντων και σημαίνει χαμηλότερη, χαμηλότερα έσοδα από τον τουρισμό και χειρότερη κίνηση κεφαλαίων. Η υποβάθμιση της ζήτησης αυτή σημαίνει για τις αφρικανικές οικονομίες απόλυτη 251 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για πολλές χώρες βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι τεράστια και φτάνουν μέχρι και την επιστημιστική κρίση. Έχουμε, αναμένεται ότι οι χώρες με λιγότερη ανάπτυξη θα έχουν ε, από 55 έως 90 εκατομμύρια πολίτες σε συνθήκες άκρας φτώχειας και αναμένεται επίσης ότι θα είναι πολύ ε, μεγάλος ο αριθμός των ατόμων που θα πληγούν από την επιστηστική κρίση. Αναμένεται ένα δισεκατομμύριο πεινασμένη στον κόσμο εφέτος. Εγώ ξεκίνησα πέρυσι την ε, Task Force ε, για τα θέματα αυτά και σας παρακαλώ να εξετάσετε και τις συστάσεις για την αντιμετώπιση των χασμάτων στις ε, δεσμεύσεις ως προς την ανάπτυξη, ως προς το χρέος, ως προς το εμπόριο και την βοήθεια. Χρειάζεται ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η κλιματολογική σταθερότητα, όπως όμως και ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, μια τάξη χρηματοπιστωτική, πρόοδο ανθρώπινη, στα θέματα των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Τα Ηνωμένα Έθνη αγωνίζονται να σταθούν στο ύψος των αναγκών. Έχουμε ένα πολύ πιο ανεπτυγμένο τώρα σύστημα διαχείρισης, διοίκησης της δικαιοσύνης και ε, λογοδοσίας, συστήματα ιστορικού ελέγχου δηλαδή, για περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και περισσότερες πληροφορίες, καταλληλότερη ενημέρωση των κρατών μερών και του κοινού. Ταυτόχρονα, την ισότητα την ενσωματώνουμε στον οργανισμό μας και έχουμε λάβει, η Γενική Συνέλευση έλαβε την απόφαση για μία ε, και μόνη ειδικά προσδορισμένη για θέματα τη ισότητα των φύλων μονάδα στα Ηνωμένα Έθνη. Πράγμα το οποίο μα διευκολύνει ιδιαίτερα ω προ την ανάπτυξη των δικαιωμάτων και τη θέση τη γυναίκα. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να πω ακόμη μερικά λόγια για το Delivering as One, την πρωτοβουλία να προσφέρουμε ω ένα, όπου σημαίνει ότι κυβερνήσει, χορηγοί, δωρητέ και ομάδε κρατών των Ηνωμένων Εθνών με νέα ενεργητικότητα, με νέα αποφασιστικότητα ε, προσφέρουν λύσεις συμφωνούν σε μεταρρυθμίσεις και επιταχύνουν την αλλαγή και το δυναμικό ε, προς το οποίο πρέπει να στραφούν τα Ηνωμένα Έθνη για ένα πιο συνεκτικό σύστημα. Έτσι λοιπόν οι εκθέσεις καταγραφής της κατάστασης που προετοιμάσαν οι κυβερνήσεις και, τα, και οι ομάδες κρατών των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι υπάρχουν ελπιδοφόρες, ε, επιτεύγματα οι χώρες ε, που είχαν την, τον πιλωτικό ρόλο, όπως και άλλες ε, χώρες, ε, βλέπουμε ότι έχουν αναπτύξει πιο συνεκτικά και εστιασμένα προγράμματα και οι ομάδες κρατών των Ηνωμένων Εθνών ανταποκρίνονται πολύ πιο αποτελεσματικά ως προς τα αιτήματα των κυβερνήσεων, δίνοντας δηλαδή ουσιαστικές απαντήσεις με μία φωνή για σημαντικά θέματα χάραξης πολιτικής. Επίσης έχουμε πολύ σημαντική εξέλιξη ως προς τους δημοσιονομικούς ε, μηχανισμούς μας με το ενιαίο ταμείο One Fund που σημαίνει εναρμόνιση της κινητοποίησης κεφαλαίων και απογραφή καταλογισμό, αν θέλετε, μεταξύ των οργανισμών των ΗΕ Εθνών, με πολύ χαμηλότερο επομένω κόστο στι συναλλαγέ και τι ε, μεταβάσει των κονδυλίων. Έτσι λοιπόν τώρα ξεκινούμε για τις πιλωτικές χώρες τις αξιολογήσεις. Η Γενική Συνέλευση έχει ζητήσει από το Γενικό Γραμματέα να προβεί στις ρυθμίσεις που χρειάζονται για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της πρωτοβουλίας προσφέρουμε, αποδίδουμε ως ένας, delivering as one. Και εγώ ε, συνεργάζομαι στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών με την ε, ομάδα αξιολόγηση των Ηνωμένων Εθνών και την ομάδα ανάπτυξη, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε αυτή την ε, προσπάθεια. Κυρίε και κύριοι, έχουμε τώρα πολύ μεγάλε προκλήσει μπροστά μα. Έχουμε συνεργασία γερή όμω, συνεργασία πολυπίκυλη και εκτεταμένη που στηρίζεται στο συντονισμό των δραστηριοτήτων διατήρηση της ειρήνης και την αποτροπή των ε, συγκρούσεων που περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή ε, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση, ανταλλαγή προσωπικού και κατάρτισης, χρηματοδότηση ε, ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων των ΗΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαβουλεύσεις για την αναπτυξιακή πολιτική. Τώρα λοιπόν η έκθεση που σας παρουσιάζω σήμερα σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε σε χώρες που μόλις έχουν αναδυθεί από μια κρίση, είτε αυτή η κρίση είναι μια φυσική καταστροφή, είτε είναι ανθρωπογενής σύγκρουση. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο περιβάλλον, που συχνά χρειάζεται επιπλέον ε, δυναμικό και πόρους να αξιοποιήσουμε είναι πολύ μεγάλες φυσικά και θέλουμε όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα να επιτύχουμε. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα την αποναρκοθέτηση, έχουμε τον περιορισμό της κυκλοφορίας των όπλων και την προστασία των ατόμων και των ομάδων κινδύνου. Έχουμε επίσης βοηθήσει πρώην μαχόμενους και όλους εκείνους που έστω και έμεσα είχαν εμπλακεί σε ένοπλες συγκρούσεις να επανέλθουν στον ομαλό βίο, να επανασυνδεθούν με το παρελθόν τους και με τις κοινότητές τους, τις κοινωνίες στις οποίες ζουν. Έχουμε τα λεγόμενα δίκτυα ασφαλείας ως προς την διασφάλιση τροφίμων, ε, υγειονομικής περίθαλψης και επιστηστικής βοήθειας για εκατομμύρια των ανθρώπων εκείνων που έχουν βρεθεί εκτεθειμένη και χωρί δίχτυ ασφαλεία, Έχουμε αγωνιστεί για να δημιουργήσουμε νέες θέσει εργασία. έχουμε αγωνιστεί για να περιορίσουμε επιδημίες Έχουμε, αγωνιστεί για να αντιμετωπίσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα στις περιοχές που μόλι βγαίνουν από μια κρίση, εκεί που πραγματικά υπάρχουν προτεραιότητε. Και επίση ε, αγωνιζόμαστε και για την ανοικοδόμηση των θεσμών, έτσι ώστε να κερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι προσπάθειε μα για την αποκατάσταση του κράτου δικαίου σημαίνουν ταυτόχρονα την ε, ε, υποστήριξη των υπηρεσιών ασφαλείας έτσι ώστε να επανασχεδιάσουν τον, να επανασχεδιάσουν αυτόν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, στο περιβάλλον δηλαδή του εκδημοκρατισμού. Ένα πολύ καλό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο τα Ηνωμένα Έθνη αμερόληπτα βοηθούν ε, την ε, Επιτροπή να αναπτύξει πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα. Έχουμε επί παραδείγματι υποστηρίξει τοπικές και εθνικές εκλογές στο Αφγανιστάν, στην περιοχή των Μεγάλων Λίμνων στην Αφρική και τη Δυτική Αφρική και έχουμε, ανα... έχουμε υποστηρίξει και τρεις ε, διαφορετικούς προεκλογικούς γύρους στο Ιράκ στην τελευταία πενταετία. Η έκθεση χωρίς να υποβιβάζει τις ε, δυσκολίες που υπάρχουν σε χώρες αναδιόμενες μόλις από μια κρίση δεν ε, μπορεί και να παραγνωρίσει την σημασία της διεθνούς υποστήριξης. Η συνεταιρική μας σχέση πάντοτε, μπορείς, πάντοτε μπορούσε και μπορεί να βελτιώνει ζωές, να περιθωριοποιεί εκείνους που προσπαθούν να ανατρέψουν την εξομάλυνση, να σταθούν εμπόδια στην εξομάλυνση και στην ειρήνη και να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξαναβρούν ελπίδα για, το, για ένα καλύτερο μέλλον. Και πέραν της ε, ανοικοδόμησης, ε, αυτό που ζητούμε είναι η, καλή, ανοικοδόμηση προς το καλύτερο, δηλαδή να μην ξαναγυρίσουμε σε προϋπάρχοντα ενδεχομένω προβλήματα. Στο Πακιστάν είναι παραδείγματι η ενισχυμένη συμμετοχή των κοριτσιών, το η παρουσία των κοριτσιών στο σχολείο και η αποκατάσταση μιας ε, κοινότητας, μιας κοινωνίας πολύ πιο βιώσιμας, βιώσιμης, σημαίνει ότι μπορούμε να αποφύγουμε κρίσεις και προβλήματα του παρελθόντος. Η εταιρική μας σχέση σημαίνει ταυτόχρονα ότι ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας είναι ρόλος υποστηρικτικός των εθνικών φορέων που τους επιτρέπει να αναλάβουν και πάλι τα ενία όταν είναι σε θέση να το πράξουν για τη δική τους ανάπτυξη. Και επίσης έχουμε αναπτύξει και τις λεγόμενες υποδομές της ειρήνης με τις διαδικασίες και τις ικανότητες που χρειάζονται οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών όπου τις χρειάζονται. Ταυτόχρονα η έκθεσή μας υποστηρίζει και επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα μιας ανεξάρτητης αξιολόγησης που είχε αναπτύχθηκε το 2008 υπό την αιγίδα της Επιτροπής και που ορίζουν ή που λένε ότι η Επιτροπή μπόρεσε χάρη στην εργασία με τα Ηνωμένα Έθνη να προσφέρει βοήθεια εκεί όπου δεν θα μπορούσε διαφορετικά να την έχει προσφέρει για την ε, ε, εμπλοκή σε περιβάλλοντα μετά την εκδήλωση κάποιας κρίσεως και ότι επίσης έχει αξιοποιήσει πολύ σημαντικά τον προνομιούχο ρόλο που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη ως προς τον διάλογο, τον ειρηνικό διάλογο με τις ε, κυβερνήσεις, τον συντονισμό που προσφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη και βέβαια και την, ε, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης στους οποίους μπόρεσε να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι χορηγοί και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε βοηθήσει στην επίλυση πολλών και λησμονημένων ακόμη κρίσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες Εμεί στα Ηνωμένα Έθνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη προσφέρει στην ε, ανάπτυξη, ε, στα προγράμματα ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια που αναπτύσσουμε σε περισσότερε από 100 χώρε, ε, τόσο στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, την ενίσχυση τη διακυβέρνηση, τι επενδύσει στην υγεία, την εκπαίδευση, τα ύδατα και τις ε, συνθήκες ε, αποχέτευσης και σας καλώ όποτε βλέπετε ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν, είναι ικανοποιητικό για σας να μιλάτε και να επισκέπτεστε τους ε, παράγοντες των ΗΠΑ που βρίσκονται στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Parlement qui la Madame Crétu l'a demandé. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στις Βρυξέλλες και που επισκεφτήκατε την Επιτροπή μας. Οι ερωτήσεις μου θα εστιαστούν στα εξή. Όπως είπατε, σημειώθηκαν πρόοδοι τον τελευταίο καιρό στην εξάλληψη της φτώχειας. Το ερώτημά μου όμως είναι το εξής. Με την οικονομική αυτή κρίση υπάρχει μία στρατηγική για τη θέση νέων προτεραιοτήτων για τις εταιρικές σχέσεις. Επίσης, εσείς μπορείτε να παροτρύνετε τις χώρες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την αναπτυξιακή βοήθεια και αναφέρομαι στο 0,7 του ΑΕΠ. Πώς μπορούμε να σπρώξουμε τις πλούσιες χώρες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Και επίσης να σας ρωτήσω για τις γυναίκες και την ανάληψη της εξουσίας από γυναίκες. Ήσασταν και υπουργό για τις γυναίκες και τα παιδιά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι γυναίκες, ιδιαίτερα στην τομέα, στην τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης, της ανάπτυξης της ειρήνης. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω και μια ερώτηση σχετικά με το μέλλον των γυναικών. Grazie Presidente, ringrazio la signora Mighiro per il suo rapporto e io credo che siamo in un periodo estremamente importante, cioè noi stiamo vedendo come Eh, c'è in Εξετάζουμε πώς θα δημιουργηθεί μια παγκόσμια κυβέρνηση. Πώς θα έχουμε και μια μεταρρύθμιση του ΟΗΕ που θα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αναφέρουμε σε αυτό το οποίο είναι μια προστακτική πλέον αναγκαιότητα, μια συμφωνία για να καταλήξουμε στην ρύθμιση της εκπομπής αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και πρέπει οπωσδήποτε αυτό να γίνει στην Κοπεχάγη. Ξέρουμε καλά ότι όλα αυτά είναι θέμα αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μία κοινή μέθοδο και μία κοινή διαχείριση. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε έναν, ε, ένα σπόρο μιας νέας παγκόσμιας διακυβέρνησης στον τομέα αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει, διότι η Ένωση η ίδια αποτελεί ένα, ένα πειραματικό εγχείρημα μιας υπερεθνικής κυβέρνησης. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμεύσει ως παράδειγμα και για την εξέλιξη των Ηνωμένων Εθνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή αυτή η μεταρρύθμιση που θα μπορέσει να εγγυηθεί και μία μεγαλύτερη συμμετοχή των λαών στη διαχείριση του ΟΗΕ, δηλαδή μία μεγαλύτερη δημοκρατική υπόσταση, έναν δημοκρατικό έλεγχο στον ΟΗΕ. Θέλουμε λοιπόν εμείς αυτή η συνεργασία να οδηγήσει και σε μία πιο προθυμένη μορφή δημοκρατίας με εμπιστοσύνη, αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία. Ο κύριος Κέσλερ Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και εγώ κυρία Δόκτωρ Μεγκύριο, ξέρω ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ σε γενικές γραμμές λειτουργεί πάρα πολύ καλά και το ξέρω από τη δική μου τη δουλειά και ότι έχω επισκεφθεί και πολλές ε, χώρες, στην Αγγόλα, τη Λατινική Αμερική. Αυτό που με απασχολεί είναι το εξή. Εσείς πώς θεωρείτε ότι η συνεργασία με τα μεμονωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αναπτυχθεί σε ό,τι αφορά την ε, μεμονωμένη πολιτική ανάπτυξης θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά συντονισμένη με τη συνολική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αξιολογείται λοιπόν τη δράση άλλων κρατών εκτός της Ένωσης στις διάφορες αναπτυσσόμενες χώρες. Είδαμε για παράδειγμα στο Ανατολικό Τιμόρ ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν χωρίς όμως να υπάρχει συντονισμός και έτσι σημαντικές διαδικασίες για την ανοικοδόμηση της χώρας ουσιαστικά παραμποδίστηκαν, παρακολούθηκαν. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα συντονισμού από τον ΟΗΕ σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει καλύτερος πραγματικά συντονισμός. Ο κύριος Σαλαφράγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ Είναι πολύ σημαντική η παρουσία της και οι επαφές μεταξύ ΟΗΕ και αυτού του κοινοβουλίου θα πρέπει να γίνονται τακτικότερα. Την καλωσορίζουμε λοιπόν ιδιαίτερα. Σε αυτή την καταπληκτική έκθεση όπου αναλυτικά αναφέρεται ποια ήταν η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών ε, και ο ΙΕ. Βλέπουμε επίσης ποιος είναι ο προϋπολογισμός, πόσο συμμετέχουν τα κράτη μας, ε, όπως επίσης και πώς συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, είπε και ο προλαλήσαντας ο προλαλήσας συγγνώμη, συμμετέχοντας ως παρατηρητή, της ε, σε διάφορες εκλογικές διαδικασίες, στο Αφγανιστάν, στο Λίβανο, μπόρεσα να, δω, να διαπιστώσω προσωπικά την ε, καλή συνεργασία μεταξύ ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα όμως, μιλώντας ε, για, ακριβώς για συνεργασία, θα ήθελα η κυρία Μιγύρο να μας πει μερικά πράγματα σχετικά με την μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Γνωρίζουμε τη θεμελιώδη χάρτα του Σαν Φρανσίσκο, ξέρουμε ότι οι, βασικοί, οι συνθήκες από τότε έχουν αλλάξει σημαντικά. Είναι πάνω από 190 χώρες που συμμετέχουν στον ΟΗΕ. Και έχει αλλάξει ιδιαίτερα ο ρόλος του ΟΗΕ μέσα από την παγκοσμιοποίηση, μέσα από τις νέες συνθήκες ε, που δημιουργήθηκαν μετά από την, ε, την κατάργηση απεικιοκρατίας. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι λέτε για τη μεταρρύθμιση για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα βέτο των μονίμων, ε, το μονίμως εδρευόντων στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θα έπρεπε να το αλλάξουμε και δεν θα έπρεπε ο... η αποτελεσματική πολυμερότητα που εμείς ε, θέλουμε στην πολιτική ε, πώς θα μπορούσε να γίνει πλέον έργο και όχι μόνο λόγια. Θα ήθελα λοιπόν να μου εξηγήσει η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας πώς έχει η μεταρρύθμιση. Δόκτωρ Μιγύρο, παρακαλώ μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ και όλους τους ε, μιλητές για, ε, για τα πολύ ευγενικά τους λόγια. Την πρώτη ερώτηση ομολογώ ότι δεν την άκουσα 100% γιατί πάλευα με τα ακουστικά μου να καταλάβω από πού θα ακούσω την ε, διερμηνία. Μου λέει τώρα ο συνάδελφος ότι η ερώτηση αναφερόταν στα μέσα που μπορεί να έχουν στη θέση του τα Έθνη έτσι ώστε να ε, πιέσουν ε, τα κράτη να διαθέσουν το 7% επί του ΑΕΠ. Αυτό που θα σας πω εγώ το είναι το εξής, ότι όποτε μπόρεσε ο Γενικός Γραμματέας μέσω της διεθνούς κοινότητας, του G8 δηλαδή, του G20, του G20 δηλαδή, ε, να μιλήσει πάντοτε επικεντρωνόταν στην ανάγκη να υποστηριχθούν αυτές οι πρωτοβουλίες, τα MDGs, που είναι και το βασικότερο μέσο που έχουμε για την ανάπτυξη. Άλλοι λοιπόν ικανοποίησαν το στόχο του 0,7% επί του ΑΕΠ, άλλοι μάλιστα το ξεπέρασαν. Καθήκον μας λοιπόν παραμένει η, ε, ο αγώνας να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ε, πιέσουμε έτσι ώστε δεσμεύσεις του Μοντερέι, του Γκλένιγκολς, του Λονδίνου να τηρηθούν. Όμως έχουμε και σημαντικές επιτυχίες να επιδείξουμε και αυτό παντα το υπενθυμίζω. Και γνωρίζουμε ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει πλήξει ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύουμε πάντως ότι εάν θέλουμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τους λοιπούς πυλώνες των Εθνών, άλλη λύση δεν υπάρχει από αυτήν. Και επίσης ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται στην υπόθεση αυτή. Ο Γενικός μας Γραμματέας ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην παρουσία των γυναικών στο Ηνωμένα Έθνη. Είχαμε από την ανάληψη των καθηκόντων του περί το 40% αύξηση του αριθμού των ε, γυναικών στο προσωπικό και 9 γυναίκες έχουν αναλάβει καθήκοντα σε ένα το επίπεδο. Έχουμε παραδείγματι επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας, μάλλον αναπληρώτρια ε, επικεφαλής. Ε, στο πρόγραμμα των Εθνών για την ανάπτυξη, το UNDP, έχουμε την κυρία Μάργκρετ Λόι, επίσης ε, ως ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέως, ειδική επεσταλμένη καλύτερα του Γενικού Γραμματέως στη Λιβερία και πολλά άλλα υψηλά καθήκοντα έχουν αναλάβει γυναίκες. Είμαστε στρατευμένοι λοιπόν στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, στην για την και συνεχίζουμε. Ταυτόχρονα όμω καλωσορίζουμε και το ψήφισμα των κρατών μελών πρόσφατα που ζητά από τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίσει μια χωριστή μονάδα για τα ε, θέματα τη ισότητα των φύλων. Πράγμα το οποίο μα λύνει τα χέρια και μα επιτρέπει να δράσουμε πολύ πιο αποφασιστικά. Δεύτερη ερώτηση. αφορούσε την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση. Και συμφωνώ με τον κύριο Βουλευτή ότι χρειάζεται η παγκόσμια διακυβέρνηση να εξυπηρετεί, να υπηρετεί καλύτερα τους μεγάλους στόχους και τις προκλήσεις εποχής. Πράγμα το οποίο επιτυγχάνουμε με τη μεταρρύθμιση των Εθνών, υπό την αιγίδα και με πρωτοβουλία του Γενικού μας Γραμματέα. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να αναφερθώ και στον κύριο Βουλευτή που αναφέρθηκε στην, στη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου ασφαλείας. Πράγμα το οποίο, όπως ξέρετε, έχει ήδη ξεκινήσει να συζητείται σε επίπεδο κρατών μελών. Το συζητούν ήδη δηλαδή το θέμα της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου, της τρόπου λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Γενικός Γραμματέας παρέλαβε πρόσβαλα πρόσφατα την ε, πρόθεσή του να συνεργαστεί ε, δραστήρια με τα κράτη-μέλη άλλα μέλη, άλλα κράτη προτιμούν χωρίς να αλλάξει το ισχύον σύστημα του δικαιώματος άρνησης να διευρυνθεί ο ρυθμός των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας ενώ άλλα κράτη θα ήθελαν να καταργηθεί το δικαίωμα άρνησης Πάντως, όπως και να είναι, εμείς συνεχίζουμε στον αγώνα αυτό και κάνουμε και τη μεταρρύθμισή μας από την πλευρά τη δική μας ως προς την αναρμόνιση των συμβάσεων που αναπτύσσουμε για το προσωπικό μας, έτσι ώστε όλοι να ε, εργάζονται υπό τις ε, ίδιες ε, συνθήκες και προσπαθούμε ταυτόχρονα και τα θέματα του περιβάλλοντος να τα αντιμετωπίζουμε μέσα από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, γιατί αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις αυτές, όπως διαπιστώσαμε, πολύ καλύτερα από, από κοινού. Αυτό είναι που μπορούμε να επιτύχουμε, να έχουμε δηλαδή πιο πολύ πολιτική βούληση, να έχουμε περισσότερη αιστεία στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κλιματολογικές αλλαγές. Βέβαια, γεγονός παραμένει ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μια συμφωνία για την παγκόσμια διακυβέρνηση και για τις κλιματικές αλλαγές. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεργαστεί πολύ μαζί μας και πολύ καλά μαζί μας. Τα κράτη-μέλη που έχουν δεσμευθεί, παραδείγματι, στην ε, μείωση των εκπομπών τους, αλλά ταυτόχρονα και η προβλέψη και ο περιορισμός των συνεπειών ε, των κλιματικών αλλαγών είναι μέσα στις προοπτικές που θα πρέπει να διερευνήσουμε ακόμη περισσότερο. Επίσης, όσον αφορά την ερώτηση τη σχετική με τη συνεργασία με επιμέρους κράτη-μέλη, εάν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Εμείς συνεργαζόμαστε μέσα από το πλαίσιο συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών. Παραμένει όμως εμφανές ότι ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν αυτός ο συντονισμός ε, φαίνεται ότι είναι σκοπιμότερο να στραφεί προς την ε, διαχείριση των πόρων μας κάποιο διαφορετικό διακόπτη μιλήτρια. Μου υπενθυμίζει εδώ ο συνάδελφος και τον ευχαριστώ ότι έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς για την ε, κατανομή εργασίας που έχει ε, του οποίου είχε την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προχωρούμε λοιπόν ακόμη περισσότερο και θέλουμε να προσδιορίσουμε ποιο αναλαμβάνει τι και έτσι να αναπτύσσουμε και τα προγράμματα που θα έχουν πολύ, καλύτερη, α, πολύ καλύτερο αντίκτυπο και ως προς την αξιοποίηση των πόρων, αλλά και ως προς τον συντονισμό και την εστίαση, τη στόχευση καλύτερα στους τομείς προτεραιότητας. Άλλη ερώτηση σε ποιο επίπεδο έχουμε φτάσει ω προ τι μεταρρυθμίσει των ΗΠΑ, πέραν του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Έχουμε μπορέσει μέχρι τώρα, και όπως είπα και νωρίτερα, να ενισχύσουμε στο βαθμό που μπορούμε το έργο της Γενικής Γραμματείας. Αναφέρθηκα επίσης στην εναρμόνιση των συμβάσεων όσον αφορά το δικό μας προσωπικό και επίσης έχουμε θεσπίσει και ένα μηχανισμό λογιστικό πιο διαφανή και ε, που μας επιτρέπει και να λογοδοτούμε εναντί των κρατών μελών και να έχουμε λογοδοσία ως προς τους σπόρους που διατίθενται. Για να βλέπουμε δηλαδή πού πηγαίνουν τα χρήματα που διαθέτουμε. Και έτσι επίσης ενισχύεται η λειτουργία της ομάδας των πολιτικών υποθέσεων, της Επιτροπής των Πολιτικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να μην έχουμε μόνο την ε, λειτουργία της ε, αποκατάστασης μετά μια κρίση ή της ανάνυψης μετά μια κρίση, αλλά να προλαμβάνουμε και να δρούμε και μεταγενέστερα ακόμη περισσότερο. Επίσης, στην ασφάλεια, την επιστηστική, στα θέματα του λοιμού, στα θέματα των φυσικών καταστροφών, ενισχύονται τα Ηνωμένα Έθνη ως φορέας πολυμερούς συνεργασίας και ως παράγοντας του νιου multilateralism, δηλαδή της νέας πολυμερούς συνεργασίας. Πολλοί βουλευτές ζήτησαν το λόγο. Θα περιορίσουμε το χρόνο μιλίας για ένα λεπτό για τις ερωτήσεις. Ο κύριος Στάνοκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και τη Δόκτωρα Μιτζήριο. Όλοι θέλουμε να τερματίσουμε το κλίμα της ατιμορρησίας που επικρατεί, αλλά η πραγματικότητα δυστυχώς είναι διαφορετική, γιατί η δικαιοσύνη πολλές φορές απαιτεί και την αμνηστία προκειμένου να υπάρξει πρόοδος. Ωστόσο, η ΟΗΕ έχει θέσει νέα πρότυπα καταγγέλλοντας τον πρόεδρο Βασίλη του Σουδάν και ως τώρα δεν μπορεί να ε, προχωρήσει αυτή η δίωξη, η παραπομπή. Τι έχει πετύχει λοιπόν ε, αυτή η απόπειρα πέρα από το να αναστατώσει τη Σουδανική κυβέρνηση. Η κυρία Κιάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα, θα ήθελα να σας ζητήσω να σχολιάσετε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που σχετίζεται με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και της του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά τις ε, δράσεις μας για την γεωργία. Όπως ξέρετε, το, η αποστολή παρατήρησης ε, στην γεωργία σταμάτησε φέτος λόγω παρέμβασης της Ρωσίας. Και ο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνταν πρώτου ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη δική σας αξιολόγηση για τη δέσμευση και της Ένωσης αλλά και του ΟΗΕ στην περιοχή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ως αποτυχία αυτή την κοινή μας δράση. και μήπως η συνεργασία μας έχει λειτουργήσει καλύτερα στο κοσυφοπαίδιο για ποιο λόγο και τι διδάγματα θα πρέπει να εξάγουμε από αυτές τις διαφορετικές εμπειρίες. Ο κύριος Κεραίρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Μιχύρο. Αμφισβητούνται οι στόχοι της χιλιετίας ως αποτέλεσμα της κρίσης και φαίνεται όμως να έχουμε ένα σενάριο υπέρ του πολυ... της πολυμερότητας και της ενίσχυσης του ΟΗΕ. Το είδαμε αυτό και με την ε, μεγάλη διάσκεψη κορυφής ε, για την ε, αλλαγή του κλίματος και με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ευκαιρία λοιπόν δεν είναι να ενισχύσουμε τον ΟΗΕ ούτως ώστε του χρόνου που θα έχουμε τη λήξη της προθεσμίας για τους στόχους ε, της ε, χιλιετίας να έχουμε πραγματικές ε, δυνατότητες αλλαγής και να έχουμε και πέντε χρόνια μπροστά μας επίσης για να ξεριζώσουμε τη φτώχεια από τον κόσμο. Η κυρία Ματέρα. Sì, Presidente, colleghi tutti, Madame Ghiro, intervengo oggi non Σήμερα κυρία Μιγύρο παίρνω το λόγο όχι για να κάνω ερώτηση αλλά για να σας ευχαριστήσω. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής ΦΑΜ δικαιώματα της ε, γυναίκας. Ε, είμαι από το ΕΛΚ και αντιπροσωπεύω την Ιταλία. Είμαι πραγματικά περήφανη που συναντώ εδώ μία γυναίκα σύμβολο για την Αφρική. Ωραία πράγματα λέτε, λέει ο πρόεδρος, πολύ ωραία πράγματα. Να, τα ξαναπώ όλα από την αρχή, λέει ο ομιλήτρια. Αν Allora, Presidente, colleghi tutti, intervengo oggi... No? να μην τα ξαναπώ από την αρχή, ξεκίνησε ο μιλητή να τα ξαναλέει από την αρχή. Είπα ότι δεν παίρνω το λόγο για να σας κάνω μια ερώτηση, αλλά για να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΦΑΜ, δηλαδή ισότητας μεταξύ, μεταξύ των φίλων. Αντιπροσωπεύω την Ιταλία και το ΕΛΚ. Είμαι περήφανη που συναντώ μια γυναίκα σύμβολο που παλεύει για τα δικαιώματα της γυναίκας στην Αφρική. Εσείς εδώ ως αναπληρωματική γραμματέας του ΟΗΕ <laughs> Λοιπόν, κυρία Μιγύρο, το βιογραφικό σας είναι πραγματικά φανταστικό. Λέει εκπληκτικά πράγματα για σας. Διότι πέρυσι όπου στο στην πρώτη συνάντηση G8 των γυναικών ήσασταν πρωταγωνίστρια εσείς ε, και υπουργό Γκαρφάνια. Eh, ε, προσπαθήσατε να εμπλέξετε και τους συναδέλφους μας εδώ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Απλά να σας ευχαριστήσω ήθελα για όλη τη δουλειά που κάνατε και που θα συνεχίσετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτηση για την παγκόσμια δικαιοδοσία και το ρόλο του παγκόσμιου του δικαστικού διεθνούς δικαστηρίου, ποινικού δικαστηρίου και το κατά πόσο υπάρχει θέμα τιμωρησία. Νομίζω ότι το γεγονό ότι υπάρχει το δικαστήριο αυτό αποτελεί σύμβολο καταδίωξη, δίωξη, αν θέλετε, των δικτατοριών. Αυτό αποτελεί από μόνο του επίτευγμα. Και η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι να συνεργαστούμε με το ICC, με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι γεγονός ότι δεν έχει αποδώσει καρπούς ακόμα ε, το θέμα της παραπομπής του Προέδρου του Σουδάν. Αλλά είτε σε περιφερειακά σώματα, είτε σε επίπεδο Διεθνούς ε, Ποινικού Δικαστηρίου υπάρχει δίωξη των εγκλημάτων. Ξέρουμε ότι στο δικαστήριο της Χάγης υπάρχει το δικαστήριο για τη Ρουάντα. Έχουμε την παραπομπή ε, ηγετών όπως του Charles Taylor. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτά τα μέσα που μας βοηθούν να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία. Αυτό που χρειάζεται είναι η συνεργασία. Και ο Γενικός Γραμματέας έχει καλέσει επανελειμμένα το Σουδάν να συνεργαστεί. Ξέρουμε ότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα στην Αφρικανική Ένωση για να αντιμετωπιστεί το θέμα, αλλά όλοι ε, αναμένουμε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας, για την ε, πρόληψη των συγκρούσεων και τις σχετικές προσπάθειες που γίνονται στη Γεωργία. Θεωρώ ότι το έργο του ΟΗΕ και η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ δεν αποτελεί αποτυχία δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία. Θεωρούμε ότι όλα τα μέρη έχουν μία υποχρέωση. Μία υποχρέωση να τηρήσουν τα όσα υποτίθεται ότι θα πρέπει να κάνουν για να τηρηθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα για τα MDGs για του χρόνου. Σωστά είπατε ότι είναι κρίσιμη η, επόμενη εποχή. Το 2010 αποτελεί ημερομηνία στόχο και ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε το Σεπτέμβριο να γίνει μια συνεδρίαση για μια αναθεώρηση, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά και για να δούμε πώς πάει η εφαρμογή των προγραμμάτων στις διάφορες, στις διάφορες χώρες. Και τα προγράμματα στην ε, Αφρική είναι αυτά τα οποία είναι τα πιο αμφιλεγόμενα. Είναι πραγματικά αναμένουν ότι θα πετύχουν τους στόχους τους τα θέμα λοιπόν εφαρμογή. Καλό λοιπόν, καλό τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, υποστηρίζουν τα MDGs, αλλά και να δραστηριοποιούνται προκειμένου να τηρούνται οι υποσχέσεις, οι δεσμεύσει για τα MDGs. Να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και θα πρέπει να συνεχίσουμε την σωστή συνεργασία προκειμένου να μην υπάρχουν μόνο λίγες γυναίκες ε, σε υψηλές θέσεις, αλλά πολλές. Και νομίζω ότι η συνεργασία μας μας την δίνει αυτή την ευκαιρία. Μιλήσαμε για τη διάσταση του φίλου και θα είναι σημαντικό να παραμείνετε δεσμευμένοι προς αυτό το σκοπό και θα χαρούμε να υποδεχτούμε τους βουλευτές που θα μας επισκεφτούν προς αυτό το σκοπό και σκοπεύουμε φυσικά να σας ενημερώσω λεπτομερώς για τα θέματα αυτά. La parole est maintenant à Monsieur Ευχαριστώ. Το λόγο και εγώ είχε ο κ. Πλεύρης, παρακαλώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και θέλω να ρωτήσω πρώτον στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που υπάρχει και με δεδομένο ότι πολλές χώρες μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις για βοήθεια των αναπτυσσομένων χωρών. Υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους στις αιστείες τους και να περιοριστεί στο μέτρο του εφικτού η μεταναστευτική ροή προς την Ευρώπη που συνεχώς αυξάνεται. Δεύτερον, για το Αφγανιστάν θέλω να σας ρωτήσω. Εάν είστε ικανοποιημένοι για την πρόοδο που υπάρχει μετά τις πρόσφατες εκλογές και επειδή ακούσαμε βέβαια πολλά να λέγονται για το ρόλο της γυναίκας και είναι θετικό αυτό, ποιε ήταν οι συγκεκριμένες ενέργειες των Ηνωμένων Εθνών για τον απαράδεκτο νόμο που υπήρξε στο Αφγανιστάν, όπου ουσιαστικά προσέβαλε την αξιοπρέπεια των γυναικών, καθώς επέτρεπε στον σύζυγο να απαγορεύει τη σύντηση κάτω από ορισμένε προποθέσει. Υπήρξαν συγκεκριμένε ενέργειε από τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ένδειξη ευχαριστειών για την παρουσία της κυρία Μιγκίτο εδώ θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Είναι με την έννοια να αξιοποιήσουμε την εδώ παρουσία της και την ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων. Θέλω να πω ότι επειδή πράγματι τα παγκόσμια προβλήματα έχουν, τα προβλήματα έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα πρέπει να ενισχυθεί ο, ο ρόλος του ΟΗΕ όπως τόνισε και η κυρία Μεγκύρο στην εισήγησή της. Η ερώτηση λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, ας μας κάνει μια αξιολόγηση, δηλαδή στην ενίσχυση της πολιτικού ρόλου του ΟΗΕ και πιο συγκεκριμένα υπάρχουν κρίσιμα ραντεβού που είναι κάτω από την αιγίδα του ΟΗΕ το επόμενο διάστημα. Τι κοπεχάει για το κλίμα, το Μάρτι για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων. Εκεί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε αυτά τα ραντεβού να έχουν επιτυχία και να βγάλουν αποτελέσματα. Και μια τελευταία ερώτηση. Στη σύμβαση, στο τρίτο κεφάλαιο προβλέπει σε εθνικό επίπεδο μέτρα για την ποινικοποίηση και την επιβολή του νόμου σε αδικήματα όπως δωροδοκία δημοσίων λειτουργών. Δωροδοκία δημοσίων λειτουργών. Εδώ τώρα υπάρχει βέβαια συνεχή... Ο κύριος Δέβα όχι, όχι, ένα λεπτό είπαμε, ένα λεπτό και άμα είναι ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ο κύριος Δέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τη δόκτωρα Μικρό για τον Βίκτορ Κόλμπρετ, επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας του ειδικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, ο οποίος ε, ε, κατήγγειλε την σε εκλογές, ότι 1500 εκλογικά κέντρα δεν είχαν ελεύθερη πρόσβαση και ότι και από ό,τι φαίνεται όταν κατέθεσε την έκθεσή του ε, κινδύνευσε, πάση περιπτώσει, με απόλυση και αν ε, δεν έγινε αυτό ακόμη μέχρι τώρα θα γίνει σύντομα. Τώρα όμως βλέπουμε ότι όντως αποδεικνύεται η νοθεία στις εκλογές του Αφγανιστάν. Ε, ενώ εντωμεταξύ εμείς διαθέτουμε στρατεύματα και θέτουμε τις ζωές των Βρετανών στρατιωτών σε κίνδυνο για να προστατεύσουμε το Αφγανιστάν. Γιατί λοιπόν απελήθη ο κύριος Κόλμπρετ. Την τελευταία ερώτηση έχει ο κύριος Βανόρντεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δόκτωρ Μιγκύρο, θα επανέλθω στο ζήτημα τη αντιμετώπιση των ε, τυραννικών, των δικτατορικών καθεστώτων, πράγμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει αρκετά αποτελεσματικά η διεθνή κοινότητα. Και εδώ θα αναφερθώ όχι μόνο στα, στο ρόλο σας ως ε, εκπρόσωπο των εθνών, αλλά και στον, ε, στα προηγούμενα καθήκοντά σας ως Υπουργού της Τανζανίας και τις θέσεις που είχατε μέσα από την Σάντακ. Τώρα εγώ είδα στο Λονδίνο εκατοντάδες ατόμων που διαμαρτύρονταν ενώπιον της Νιγηριανής πρεσβείας και ιστούσαν από την Σάντο από ε, τη Ζιμπάμπουε, συγγνώμη, και από τη Σάντοκ να αναλάβει μέτρα για τον εκδημοκρατισμό στη Ζιμπάμπουε. Γιατί λοιπόν το Μουγκάμπε, το μεγάλο αυτόν δικτάτορα και τύρανο, δεν τον έχουν ελέγξει η διεθνή κοινότητα πρώτα απ' όλα, αλλά και τα γειτονικά αφρικανικά κράτη που θα μπορούσαν μη τι άλλο να υποστηρίξουν του ε, πολίτε τη Ζιμπάμπουε στην αναπροσπάθεια για ανατροπή αυτού του δικτάτορα. Ο κύριο Νέβα υπεστήριξε. Ευχαριστώ τώρα η Επιτροπή την οποία εκπροσωπεί και ο, ο, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΤΚΟ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε και εμείς δύο λόγια, κυρία Πρόεδρα, Η κυρία Μαγκύρο ε, έχει επισκεφθεί δύο επιτρόπους της, κυρία Φρελνό Βάρντεν και τον κύριο Ντεχούχτ. Ακτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η παριθμόν δύο του ΟΗΕ ήρθε στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει αυτή την έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΗΕ. Όντως, η συνεργασία ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντική σε οικονομικούς όρους. 1,2 δισεκατομμύρια το 2008 περίπου, 676 εκατομμύρια για ανάπτυξη και περίπου 400 για την ανακούφιση σε περιπτώσεις ε, έκτακτης ανάγκης. Αλλά πέρα από αυτό το στοιχείο εκτιμούμε και τις πτυχές που υπερβαίνουν το οικονομικό ζήτημα. Οι πολιτικές μπορεί να μην ε, έχουν ως πάντα αποτελέσματα συμβάσεις, αλλά πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικές και όταν προάγουμε θέματα όπως το φύλλο, η προστασία του κλίματος, καταφέρουμε να μεταδώσουμε ένα πιο ισχυρό μήνυμα από κοινού από ότι ο καθένας μόνος του. Άρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που αυτή η τέταρτη ετήσια έκθεση έχει πλέον καταστεί μια πολύ αναλυτική και αξιόπιστη έκθεση. Και ήδη η πρώτη έκθεση με την καταγραφή της κοινή μας προσπάθειας ήταν μια πολύ σημαντική προσπάθεια και την εξετάσαμε με πολύ προσοχή. Ωστόσο η έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνει και θέματα πολιτικής συνεργασίας. Η περσινή ανεξάρτητη έκθεση κατέδειξε ότι ο ΟΗΕ έχει ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη σε καταστάσεις άμεσης κρίσης και όπως τονίζεται στην έκθεση, ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι μοναδικοί πολυμερείς παράγοντες φορείς που μπορούν να παρεμβούν σε όλες τις ε, φάσεις ε, μιας κρίσης από την ανοικοδόμηση μέχρι την ανάπτυξη των κοινωνιών προκειμένου να αποτρέψουν, να προβλέψουν κρίσεις. Επίσης, η έκθεση είναι σαφής ότι με την συνεργασία μας πετύχουμε πολύ πιο πολλά από ότι ο καθένας μόνος του η υποστήριξη για παράδειγμα των αγροτών εξαρτάται και από την αξιολόγηση που γίνεται και από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμείναμε στο πλαίσιο της διατροφικής ε, και της επιστημικής ασφάλειας να συμπεριληφθούν όλες οι οργανώσεις ε, του ΟΗΕ. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας μηχανισμός ε, συντονισμού υπό τον επικεφαλής David Navarro, τον υποδιευθυντή της, Ευρωπαϊκής, ε, της Επιτροπή. Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα η συνεργασία μας λοιπόν αυτή ενθαρρύνεται και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η αντίδραση στον κύκλο Νάιτζελ ήταν ε, αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών για να αντιμετωπιστούν τα σύνθετα πολύπλοκα ζητήματα πολιτικής φύσεως που προκύπτουν στην Μιανμάρ και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα όπως το Ιράν, το Σουδάν, η Γεωργία και το καθεξής. Επίσης, ε, αυτή η έκθεση είναι πολύ ευδιάκριτη και ε, περιλαμβάνει το στοιχείο της λογοδοσίας. Είναι μια πολύ δυναμική ανακοίνωση που ε, κοιτάει, αν θέλετε, τη συνεργασία με ολιστικό, συνολικό τρόπο, προκειμένου να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της συνεργασία μας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο της ε, λογοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την έκθεση. Καταδεικνύει λοιπόν η έκθεση αυτή με πραγματικό τρόπο πώς ε, τα οι κοινωτικοί πόροι ε, συνεισέφεραν για να ανανεωθεί η ελπίδα, για να προστατευτούν οι ζωές προσπαθούμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερα από τη συνεργασία μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρουμε γιατί και πότε συνεργαζόμαστε, αξιολογώντας με κριτικό πνεύμα όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Το Κοινοβούλιο άσκησε κριτική για το ότι δεν ήταν πάντα σαφές γιατί επιλέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εταίρος. Απαντήσαμε με μια σχετική αξιολόγηση πρόσφατα όπου αναφέραμε τις καλύτερες περιπτώσεις συνεργασίας. Και η Επιτροπή λοιπόν και ο ΙΕ θα πρέπει να εξετάσουν τις δυνατότητες συνεργασίας περαιτέρω. Και ένα τομέα όπου αποδείχθηκε ότι η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή ήταν σε περιπτώσεις μετά από σε περιπτώσεις ε, ανοικοδόμησης. Θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι αρχές να συντηρηθούν σε υψηλό επίπεδο. Ακόμα και όλες οι δωρητρίες χώρες ε, αποφασίσουν να αφιερώσουν το ίδιο ποσοστό, μπορεί να αποδειχθεί ότι τα ποσά και οι πόροι που αφιερώνονται για την αναπτυξιακή βοήθεια δεν επαρκούν. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προς όλες τις δωρετρίες χώρες. Και τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω το μεγάλο συμφέρον που έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποψηφιότητα και την ε, θέση αναπληρωτή γραμματέα για θέματα φύλου. Ελπίζουμε σύντομα να διοριστεί αυτός ο γραμματέας προκειμένου να κινητοποιήσει την προσοχή όλων εντός του, ευρωπαϊκού, εντός του συστήματος του ΟΗΕ για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ την κυρία Γενική Γραμματέα να λάβει το λόγο για να απαντήσει στις τελευταίες ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτηση σχετική με την οικονομική κρίση και το γεγονό ότι πολλές χώρες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να ικανοποιήσουν τους στόχους ανάπτυξης. Είναι βέβαια πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα η χρηματοπιστωτική κρίση δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα ταχαίως να ε, ε, κινητοποιηθούν κονδύλια. Αν δούμε πόσα κονδύλια κινητοποιήθηκαν τόσο γρήγορα για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθίσατε σαφές ότι μπορούμε, αν θέλουμε, να ε, υλοποιήσουμε τουλάχιστον κάποιες από τις υποσχέσεις μας. Αυτό λοιπόν το οποίο πάντοτε ε, υπογραμμίζει ο Γενικός Γραμματέα κ. Μπανκιμούν είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες προσπαθούν να εισαγάγουν τις ε, σωστές πολιτικές, ε, κάνουν τις προσπάθειές τους και έρχεται τώρα πια η στιγμή όπου θα πρέπει παραχρήμα να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν να ξαναπέσουν στη φτώχεια εκατομμύρια πολιτών. Αυτό που μας δείχνει η κρίση είναι ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα παράθυρο ευκαιρίας, εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση και η δραστηριοποίηση, η κινητοποίηση. Για το Αφγανιστάν. Είναι απαράδεκτο η αξιοπρέπεια των γυναικών να προσβάλλεται κατά τον τρόπο με τον οποίο προσβάλλεται στο Αφγανιστάν. Ο Γενικός Γραμματέας ε, μίλησε απερίφραστα και είπε ότι δεν είναι ανεκτή τέτοια κατάσταση. Τα Ηνωμένα Έθνη, η διεθνή κοινότητα έχουν μπροστά τους μια τεράστια πρόκληση και θα πρέπει να βοηθήσουν τη χώρα αυτή να αναπτύξει θεσμούς που θα επιτρέπουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δι των δικαιωμάτων της γυναίκας, θεσμούς ε, χρηστής διακυβέρνησης και ισότητας μεταξύ των πολιτών. Τα διεθνή προβλήματα. Ναι, βεβαίω, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σημαντικό ρόλο και πολιτικό ρόλο να διαδραματίσουν. Ταυτόχρονα όμω μπορούν και να δρούν ω διαμεσολαβητή για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων. Εσεί μιλήσατε για τα ε, για τις κλιματικές αλλαγές, ε, την αποτροπή της διάδοσης των ε, πυρηνικών όπλων και την πάταξη της διαφθοράς. Δημερώ στις συνομιλίες μου με την κυρία Πρόεδρο κατέστη σαφές ότι εάν θελούσαν οι χώρες να συνεργαστούν Προ το στόχο της οικονομικής ανάπτυξης, ένα από τα προβλήματα που θα βρουν μπροστά του είναι η διαφθορά. Ευχαριστώ δε ιδιαίτερα για την, για την υποστήριξη που μας προσφέρατε στον αγώνα και τη συνεργασία με πολλέ χώρες συμπεριλαμβανομένης ευτυχώ και της δικής μου πατρίδας Τανζανία. Για τον κύριο Κόλμπριθ. Θα πρέπει να πούμε καταρχάς για τη σχετική ερώτηση ότι τα Ηνωμένα Έθνη όπως είπε ο κύριος Σκάι Άιντε, αναγνωρίζουν όντως την οφία στις εκλογές του Αφγανιστάν. Ο κύριος Κόλμπρετ ε, επεσήμανε αυτό που, είχε που είπε ακόμη χτες στην συνέντευξη που ο κύριος Σκάι Άιντε, το θέμα είναι τα Ηνωμένα Έθνη τι ρόλο διαδραματίζουν στο Αφγανιστάν. Τι ρόλο είχαν να διαδραματίσουν στο Αφγανιστάν. Τα Ηνωμένα Έθνη είχαν ρόλο να υποστηρίξουν την την εκλογική δηλαδή διαδικασία. Όχι όμω ταυτόχρονα και να διαδραματίσουν το ρόλο του παρατηρητή στι εκλογέ. Εκεί ήταν η διαφορά. Ο Γενικό Γραμματέα, λοιπόν θεώρησε ότι για να προστατέψει την ακαιρεότητα τη αποστολή ήταν απαραίτητο να ανακαλέσει τον κύριο Κόλμπριθ δεν ήταν ζήτημα συγκάλυψης. Αυτό ακριβώς που σας λέω έγινε. Όταν, έγινε ο κύριος, όταν ε, ήρθε λοιπόν ο κύριος Σκάι Άιντι χθες για τη συνέντευξη τύπου ήταν και ο κύριος Κόλμπριθ παρόν και τον υποστήριξαν όλοι για τους ε, δικτάτορες για τα δικτατορικά καθεστώτα. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι η τελευταία οργάνωση που θα μπορούσε να ανεχθεί δικτατορικό καθεστώς και τυραννικό ε, ηγέτη. Και μάλιστα θα θυμάστε ότι και εγώ από την ε, συνεδρίαση με την Αφρικανική Ένωση είχα καταστήσει απόλυτα σαφές ότι έχει έρθει πια η ώρα να πατάξουμε τα τυραννικά και δικτατορικά καθεστώτα. Ίσως κινδύνεψε κάποια στιγμή η Αφρικανική Ένωση να αποτύχει στην προσπάθεια αυτή. Όμως τη στήριξε η Διεθνής Κοινότητα, όμως τη στήριξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χάρη σε εσά, χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να πούμε ότι επιτύχαμε αρκετά. Και αν μείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές της, τότε μπορούμε όντως να ε, καταρρύψουμε τα δικτατορικά καθεστώτα στον κόσμο ολόκληρο. Και επίση σε αυτό πιστεύω συμφωνεί μαζί μου και ο Γενικό Διευθυντή που μίλησε νωρίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ασφαλώ χρειάζεται να επιμένουμε περισσότερο στον τομέα αυτών και να βρούμε και άλλου τρόπου ενδυνάμωση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Νίγκυρο για το ενδιαφέρον της, για το πάθος με το οποίο ασχολείται με τα θέματα αυτά που μας παρουσίασε την έκθεση ήρθε εδώ να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι ε, κατέστη απόλυτα σαφές σήμερα μέσω της έκθεσης αλλά και μέσω των συζητήσεων ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού και Ηνωμένων Εθνών είναι όσο ποτέ απαραίτητη. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας. Η κυρία Μίγκυρο μας υπέδειξε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση κοστίζει στην Αφρική 261 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,6 φορές δηλαδή το ποσό που συνολικά προσφέρουμε τη σκληριακή βοήθεια η διεθνή κοινότητα ολόκληρη. Δυόμιση φορές. Μέταξυ λοιπόν ε, αυτών των μεγάλων προκλήσεων του λοιμού, της πείνας, στην οποία είναι εκτεθειμένα εκατομμύρια ανθρώπων, τι ανάγκε για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την ανάγκη για μια νέα στρατηγική και του περιορισμένου πόρου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, η συνεργασία μεταξύ μα είναι όσο ποτέ απαραίτητη. Ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα και βεβαίως ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες σας τους συναδέλφους βουλευτές που ήρθατε στη συνεδρία σήμερα. Και κύριε το πέρα στη συνεδρία σας. Ευχαριστώ.